So, ladies and gentlemen, uh, we are going to... Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε μία συναρπαστική συνεδρίαση σε ό,τι αφορά τους ευελευτές στην εκλογική παρατήρηση. Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε. Νίκολα. So, uh, it's my pleasure on behalf of the... Είναι μεγάλη μου χαρά που έχουμε εδώ μαζί μας ε, ε, τους συγκεκριμένους ομιλητές. θα ευχαριστώ και όλους ε, όσοι συμμετέχετε στην, στην διάσκεψη φιλού Λουπιπέδου. Τώρα θέλουμε να γίνει μία επικοδομητική συζήτηση για το θέμα του ρόλου και των βέλτιστων πρακτικών της εκλογικής παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένου και ενός κώδικα διοντολογίας. Οι βουλευτέ συχνά συμμετέχουν σε αποστολέ εκλογική παρατήρηση και πολύ συχνά στο πλαίσιο περιφερειακών οργανώσεων. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΣΑ, ΝΑΤΟ, Συμβούλιο τη Ευρώπη, την Οργάνωση των Κρατών τη Αμερική, ε, την Διεθνή Οργάνωση ε, Γαλοφωνίας και το καθεξής. Συμμετέχουν εκεί λοιπόν άτομα, ε, η συμμετοχή μάλλον των βουλευτών που έχουν αυτή την τεχνογνωσία και εμπειρία αυξάνει την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας. Και έχουν βέβαια και τις συστάσεις που παρουσιάζεται εκ των υστέρων υπάρχει μια διαφοροποίηση και πολυμορφία στο πολιτικό υπόβαθρο και στις απόψεις των βουλευτών και αυτό ενισχύει την αμεροληψία και ανεξαρτησία των συμπερασμάτων και συστάσεων που προκύπτουν από την εκλογική παρατήρηση. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι βασικές αρχές δεν πληρούνται όπως πρέπει σε ό,τι αφορά την αυστηρή αμεροληψία, την μη παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία, ε, το μη σχολιασμό και το καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα ζητήματα που ανακύπτουν τα τελευταία χρόνια για παραπτώματα, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών. Μπορεί να πρόκειται για δημόσια σχόλια εκτός του πλαισίου της αποστολής ή ε, να αντιβαίνουν στα πορίσματα ή ακόμα και να ε, ταξιδεύουν εκτός ε, του τόπου της αποστολής ή ακόμα και σε μη αναγνωρισμένες οντότητες. Υπάρχει μακρύς ε, κατάλογος, απλώς αναφέρομαι σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, από οικονομικής, πολιτικής ή άλλης άποψης και παραμένουν πρόβλημα. Τέτοιου είδου συμπεριφορέ λοιπόν αντιβαίνουν στι βασικέ αρχέ των διεθνών εκλογικών αποστολών και μπορούν να ε, ζημιώσουν τις σχέσεις ε, για την αξιοπιστία αυτών των χωρών. Η αξιοπιστία λοιπόν στην εκλογική, της εκλογικής διαδικασίας μπορεί να ζημιωθεί. Να σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα. Τώρα το Κοινοβούλιο πρόσφατα έχει αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα αφορούν εκλογές ε, της ανατολικής γειτονίας. Πιο συγκεκριμένα Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν. Ήταν μια ξεκάθαρη απόφαση. Τα μέλη αφενός ε, ε, αποκλείστηκαν από την αποστολή. Στην άλλη περίπτωση υπήρξε απαγόρευση για οποιαδήποτε συμμετοχή σε επίσημη αποστολή μέχρι το τέλος της ε, νομοθετικής περίοδου, της κυριοβουλευτικής περίοδου. Υπήρξαν λοιπόν συνέπειες ε, για αυτές τις ε, συμπεριφορές. Όπως περιτά για κατάλληλα σχόλια ε, δημοσίω ε, και μη τήρηση τη αρχή τη αμεροληψία και δικαιωματικότητα. Πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτού του κανόνε με τον πιο αυστηρό και εύρωστο δυνατό τρόπο. Γιατί ε, το εργαλείο αυτό είναι πραγματικά ε, αναντικατάστατο για την προώθηση ε, των βέλτιστων αυτών πρακτικών. Οι κοινοβουλευτικέ συνελεύσει ε, που παρακολουθούν τις εκλογές στον χώρο ΩΣΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κοινοβουλευτική ε, Σύνοδος ε, του ΩΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, έχουν ξεχωριστούς κώδικες ε. Και τώρα έχουμε δημιουργήσει μια, έναν κοινό κώδικα, ο οποίος τώρα υιοθετείται, έχει υιοθετηθεί και από τις τέσσερις, τα τέσσερα σώματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ε, Σύνοδος ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, έχουν εθετήσει τον κώδικα τεντολογίας και επί το περιεχομένου στα άλλα δύο σώματα. Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν καλωσορίζω τους ομιλητές μας. Έχουμε την κυρία Ιζαμπέλ Σάντος, Αντιπρόεδρος τη Κοινοβουλευτικής Συνόδου του ΟΣΑ, τον κύριο Μάριο Γκαλέα, μέλος του Κοινοβουλίου της Μάλτας, τον κύριο Όλιβερ Κάσκ, δικαστή, και μέλος της Επιτροπής της Βενετίας και την κυρία Ίγκεμπορ Ναντότηρ, που είναι Διευθύντρια της Υπηρεσίας Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Όλοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση που θα μοιραστούν μαζί μας σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στους ομιλητές για να μας μιλήσουν πιο συγκεκριμένα και για τη σημασία ενός κώδικα δεντολογίας για τους διεθνείς παρατηρητές. Για παράδειγμα, θα δούμε τα καλύτερα μέσα για την συμφιλίωση της ελευθερίας έκφρασης και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από το καθεστώ του Διεθνού Παρατηρητή. Επίση, θα ήθελα να σταθείτε και στην ε, σημασία των βουλευτών ή μάλλον τη σημασία ενό ε, μονίμου σώματος που θα απαρτίζεται από βουλευτές που θα παρακολουθεί τις εκλογικές αναμετρήσεις και θα επιβάλλει την εφαρμογή ενός κώδικα δεντολογίας, θα έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη να αναλαμβάνει δράση σε περίπτωση τέτοιων παραπτωμάτων. Έχουμε μια τέτοια δομή ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το σκοπό, το λεγόμενο DEG. Τώρα, επειδή ο χρόνος πιέζει, και για να αφήσουμε και το απαραίτητο χρονικό περιθώριο αλληλεπίδραση με τους ομιλητές. Θα ήθελα οι ομιλητές ε, να μην υπερβούν τα 5-6 λεπτά έκαστος για να υπάρξει διάλογος. Το λόγο έχει η κυρία Σιάντες. Παρακαλώ. Very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια προς ε, τους ε, διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Ε, που εξετάζει τόσο σημαντικά ζητήματα. Από το 1993 έχει ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα που για πρώτη φορά υπήρξε αποστολή για μια εκλογική αναμετρήση στην Ρωσική Ομοσπονδία. Από τότε έχουμε κάνει 116 ε, τέτοιες εκλογικές αποστολές σε 31 χώρες 50 ε, παρατηρητές τα τελευταία χρόνια και συστηματικά ε, στέλνουμε αποστολές και σε παγιωμένες δημοκρατίες και σε αναδιόμενες. Αυτό μας δείχνει ότι οι αποστολές εκλογικής παρατήρησης δεν θα πρέπει να θα πρέπει μάλλον να θεωρούνται ως μια ε, ευκαιρία ενίσχυσης των δημοκρατιών. η εκλογική παρατήρηση ενισχύει τις δημοκρατικές διαδικασίες. Όπως είπε χθε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χθες, είναι απολύτως φυσιολογικό των αποστολών παρατήρησης να ηγούνται όσοι έχουν πραγματική γνώση εκλογικών αναμετρήσεων εφόσον έχουν εκλεγεί οι ίδιοι. Θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω συντομία τις διαδικασίες μας ε, και τα, μετά τα συστήματα που άπτονται του κώδικα δεντολογίας. Έχουμε λοιπόν πάνω από 115 αποστολές με πάνω από 5.000 ε, κοινοβουλευτικούς παρατηρητές. Και έτσι κατανοείται ότι έχουμε ε, αναπτύξει πολύ συγκεκριμένε πρακτικέ και διαδικασίε. Δεν θέλω να τα παρουσιάσω σε αλλά να σταθώ σε μερικά βασικά ζητήματα που μπορούν να σα ενδιαφέρουν. Πρώτον, οι επικεφαλεί των αποστολών μα επιλέγονται από τον Πρόεδρο τη Κοινοβουλευτική Συνόδου. Και συνήθως επιλέγεται και ένας ειδικός συντονιστής. ο οποίος λογοδοτεί και στην ε, Ολομέλεια και στον Πρόεδρο της SCPA. Και αυτές οι διαδικασίες ε, πραγματικά είναι πολύ ωφέλιμες. Έχουμε επίσημους κινδύνους και επιπρόσθετες αρχές που μεταξύ άλλων είναι να μην προέρχεται κανείς από μια γειτονική χώρα ή από χώρα που έχει προβληματικές σχέσεις. Να μην είναι μέλος μιας δεμερούς ομάδας φιλίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ή να έχει άλλες, ε, άλλου είδους σχέσεις ή ιστορικό υπόβαθρο που να περιπλέγουν τα πράγματα. Και λαμβάνονται υπόψη και η διάσταση του φίλου. Έχουμε περίπου τον αριθμό των παρατηρητών στο 10% της συνολικής σύνθεσης. Αυτός είναι αποτελεσματικός τρόπος να διασφαλίσουμε ότι καμία χώρα δεν θα μπορεί να επηρεάσει εξωτερικά την ε, αποστολή μας. Τρίτον, για κάθε επιμέρους ε, αποστολή, όλοι οι παρατηρητές μας πρέπει να υπογράψουν και να επιστρέψουν στη γραμματεία ένα ε, κώδικα δοντολογίας. Και έτσι πιστοποιούν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στην περίπτωσή τους, ε, οικονομικής, πολιτικής ή άλλης φύσεως, που υποσκάπτει τη δυνατότητά τους να είναι ανεξάρτητοι παρατηρητές. Και αυτός ο κώδικας ισχύει για όλους φυσικά. Από τους 5.000 παρατηρητές και τις 170 αποστολές, μόνο τρεις περιπτώσεις είχαμε όπου έπρεπε κάποιος ε, να αποκλειστεί από μία ε, αποστολή για λόγους ε, συμπεριφοράς που δεν ήταν συμβατή με τον κώδικα τοντολογίας. Πριν από μερικούς μήνες υιοθετήσαμε την τελευταία μας διακήρυξη στο Βερολίνο και εκεί ξεκαθαρίζουμε τη διάδοση των παράλληλων ε, θεσμικών οργάνων και μιλούμε συγκεκριμένα ότι τα εθνικά, τα εθνικά κοινοβούλια δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε εκλογικές αναμετρήσεις που δεν βασίζονται σε καλά οργανωμένες και διαφανείς διαδικασίες. Ναι, συστηματική μεθοδολογία Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα είναι πολύ ψηλά ε, στις προτεραιότητές μας. Λοιπόν, υπάρχουν, υπάρχει και το φαινόμενο βέβαια ε, των ψευδών ή και των ανυπάκων, αν θέλετε, ε, παρατηρητών. Πρόκειται λοιπόν για παρατηρητές ε, που ε, ταξιδεύουν προς μια χώρα εκτός του πλαισίου των παρατηρητών. Σαφώς και δεν πρόκειται για παρατηρητές OCPA, αλλά αναφέρονται έτσι από τα λιγότερα αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης. Όμως δεν υπάρχουν μηχανισμοί κυρώσεων κατά αυτών των μερών. Όμως πρέπει να ληφθούν τέτοιου είδου δράσεις υπόψη στο μέλλον. Για τεχνικούς λόγους έχουμε περιορίσει τις, ε, τους μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων. Αλλά δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υιοθετηθούν τέτοιοι μηχανισμοί στο μέλλον για το δεύτερο ζήτημα των ε, ψευδών παρατηρητών, που συνήθως ε, είναι κάτι το οποίο στείνεται από τις ε, κυβερνήσεις για να υπάρχουν οι φύλλα προσκύμενοι προς εκείνες παρατηρητές εντός εισαγωγικών είναι μια πρακτική. Μάλιστα πέρυσι ένας συνάδελφος είδε και ένα τιμοκατάλογο υπηρεσιών. Σαν OCPA λοιπόν υπάρχει ένα σαφές μήνυμα ότι οι επισκέψεις ε, κατόπιν πρόσκληση των κρατικών αρχών δεν ισοδυναμούν με μια διεθνή αποστολή που προκύπτει από εντολή διεθνούς οργανισμού, όπως ο ΕΣΥ. Και κλείνω την παρέμβασή μου Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω, περιμένω όμως ε, το διάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τρομερά ενδιαφέρον αυτό και πάρα πολύ σημαντικό και οι κακές, ε, οι, οι, ψευδοπαρατηρητές, ε, κακές συμπεριφορές κτλ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκαλέα. Παρακαλώ κύριε Γκαλέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παρατήρηση των εκλογών έχει γίνει ε, πραγματικά ένας τομέας ε, αυτόνομος με πολλούς συγκεκριμένους κανόνες ε, που λαμβάνει υπόψη διεθνή πρότυπα και διεθνή νομοθεσία. Και τέλος ο ίδιος ο λαός όμως παραμένει αυτός ο οποίος νομιμοποιεί τις εκλογές και την αγγλική διαδικασία. Η παρουσία διεθνών παρατηρήσεων μπορεί να αποτρέψει τη διαφθορά, την ε, ψήφο, την, λαθροχειρία ε, και την, να προωθήσει την δημοκρατία. Ε, και βεβαίως γενικό στόχο έχουν οι αποστολές αυτές την εν γέννη βελτίωση των εκλογικών διαδικασιών. Η παρατήρηση, παρακολούθηση των εκλογών βασίζεται στις δημοκρατικές αρχές, την ενισχυμένη δημοκρατία, το δικαίωμα του εκλέγει και το εκλέγεστε ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ε, και μαζί με αυτά την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία του εκφράζεστε, την ελευθερία κυκλοφορίας, οπωσδήποτε διαδικασία χωρίς διακρίσεις και διακριτικές μεταχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό και εμείς ως βουλευτές μπορούμε να παρατηρήσουμε εκλογές με τον πιο αντικειμενικό τρόπο. Ε, είναι γεγονός ότι στη διάρκεια της παρατήρησης των εκλογών ε, την χάνουμε ε, ε, καλής αντιμετώπισης ε, από, τις, από τους εμπλεκόμενους στις εκλογές, διασφαλίζοντας και την ακαιρεότητα της διαδικασίας. Υπήρξε και ένα σκάνδαλο όσον αφορά παρατήρηση εκλογών από το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, στο Αζερμπαϊτζάν συγκεκριμένα. Ε, ήταν ε, πολύ συγκεκριμένα τα προβλήματα της εκλογικής αυτής διαδικασίας, κυρίως δε όσον αφορά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως, ο επικεφαλής της αποστολής έδωσε πράσινο φως σε αυτές τις ε, ε, εκλογές δηλώνοντας με σοκαριστικό τρόπο ότι ήταν μια εκλογική διαδικασία ε, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εμείς μελετή, εγώ μελέτησα το θέμα αυτό μέσω μιας μέσω ενός εγγράφου το οποίο ονόμασα Caviar Diplomacy, διπλωματία του χαβιαριού, ε, διότι το, συνήθ, σύνηθες ε, δώρο της, ε, του Αζερμπαϊτζάν σε αυτές τις αντιπροσωπίες ήταν δύο κιλά χαβιάρι, τα οποία είναι της καλύτερης ποιότητας και άλλα δώρα όμως όπως μεταξωτά χαλιά και δωρεάν διακοπές κτλ. Ο επικεφαλής της ο, ο, ο Επιτροπής ε, παρατηρήσεις μαζί με ε, δύο άλλους βουλευτές, με δυστυχώς ένας εκ των οποίων ήταν από τη Μάλτα, ε, είπαν ότι οι εκλογές ήταν μια χαρά. Ωστόσο, ε, ε, ωστόσο εμείς ε, είπαμε ότι αυτές οι εκλογές ήταν πολιτικό θέατρο και οι διεθνείς παρατηρητές έπαιξαν το παιχνίδι των κομπάρσων σε αυτήν την διαδικασία. Βεβαίως είναι γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση όπως και σε άλλες περιπτώσεις η διαφθορά ήταν πάρα πολύ, έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και απέτρεψαν την σωστή εργασία της ομάδας παρατήρησης. Μας ενδιαφέρει λοιπόν, λοιπόν ε, η ε, σωστή, αδέκαστη παρατήρηση εκλογών. Ε, Από την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα εκλογές οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε πλαίσια μη δημοκρατίας, σε πλαίσια αίματος και βίας. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές θα ήταν πολύ χειρότερες εκλογικές διαδικασίες αν δεν υπήρχαν οι παρατηρητές των εκλογών. Ε, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα εθνικά κοινοβούλια τα οποία επιλέγουν ε, τις, ε, τα μέλη που θα συμμετάσχουν σε επιτροπές παρακολούθησης έχουν μεγάλη ευθύνη. Πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιωθούν ότι ο επιλεγής βουλευτής θα αποτελεί asset και όχι liability για τις εκλογικές διαδικασίες. Βεβαίως και εδώ είναι μια ιστορία που αφορά μεμονωμένα άτομα ά. Ε, και ε, επομένως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πιστεύω ότι ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί στα πλαίσια και της, του, της, Συμβουλίου της Ευρώπης μια, ένας κώδικας καλών πρακτικών που θα είναι δεσμευτικός για τους συμμετέχοντες βουλευτές στο έγγραφο το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως. Αυτά τα λέω αναλυτικά οι βουλευτές οι οποίοι συμμετέχουν σε επιτροπές παρακολούθησης ε, θα πρέπει να είναι ε, αδέκαστοι, να έχουν ε, ακαιρεότητα, να έχουν επαγγελματική συνείδηση και συνειδησιακή ανεξαρτησία. I Τελειώνοντας μπορώ να πω ότι επί δεκαετίες η παρατήρηση εκλογών έχει προωθήσει ε, την ε, δημοκρατία και έχει βοηθήσει τους ε, πολίτες. Το μέλλον τώρα τον, της παρατήρησης εκλογών εξαρτάται από μας. Πρέπει να το προστατέψουμε το δικαίωμα αυτό και να αγωνιστούμε έτσι ώστε να το βελτιώσουμε. Αλλά βεβαίως να μην λησμονούμε ότι η πρώτη δέσμευσή μας είναι η ακαιρεότητα και η ανεξαρτησία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Τηρήσατε και τον χρόνο που σας έδωσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν που θίξατε το πολύ προβληματικό αυτό θέμα της διπλωματίας του Χαβιαριού. Νομίζω ότι όλοι έχουμε παρόμοιες εμπειρίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τώρα να έρθουμε στην Επιτροπή της Βενετίας και να ακούσουμε τον κύριο Όλιβερ Κάσκ, δικαστή και μέλος της Επιτροπής της Βενετίας. Ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πολύ ενδιαφέρουσα διάσκεψη σήμερα. Καταρχάς, να εξηγήσω λίγο ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής της Βενετίας, την οποία ίσως τη γνωρίζετε από τις νομοδοτήσεις ε, για την ε, ε, Ουγγρική νομοθεσία για τα ΜΜΕ, και τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, στον ε, δικαστικό κλάδο. Η Επιτροπή της Βενετίας είναι Επιτροπή για την εδραίωση της Δημοκρατίας μέσω του, της νομοθεσίας και έχει τον στόχο να αξιολογεί την νομοθεσία στο στεγματικό δίκαιο. διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ στεγματικών δικαστηρίων και στεγματολόγων στα κράτη-μέλη που αποτελούν μέλη της για τον εκλογικό νόμο τώρα, οργανώνουμε κάποιες διασκέψεις ε, ετησίως για την ε, ε, εκλογική παρατήρηση. Φέτος έγινε στο Όσλο για την ασφάλεια των εκλογών, ήταν το θέμα. Έχουμε έναν κώδικα ε, καλών πρακτικών για τα εκλογικά θέματα. Είναι αρκετά παλιό το έγγραφο αυτό, το 2002 υιοθετήθηκε. Και από τότε έχουμε υιοθετήσει διάφορε κατευθυντήρε γραμμέ, εκθέσει για διάφορα θέματα που άπτονται τη εκλογική νομοθεσία, α πούμε, αντιμετώπιση τη ε, κατάχρηση των ε, διοικητικών πόρων κατά τη διάρκεια των εκλογικών εκστρατιών, ή ε, περιορισμούς ε, του εκλογικού σώματος, ε, τα θέματα των κατοφλίων στις εκλογές κτλ. Επίσης έχουμε βοηθήσει την κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στην, στις αποστολές εκλογικής παρατήρησης από το 2004 και έπειτα. Έχουμε λοιπόν αρκετά μεγάλη εμπειρία. Ε, knowledge about... και γνώση φυσικά για τις πραγματικές εκλογές. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι αυτή στην οποία εκφράζονται τα περισσότερα προβλήματα για θέματα εκλογών. Είναι δύσκολο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ε, διεθνή παρατήρηση εκλογών όταν ε, προκύπτουν ε, περιπτώσεις διπλωματίας του χαβιαριού ή, όπως, ή περιπτώσεις όπως αναφέρθηκαν πριν στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Η κοινοβουλευτική συνέλευση τον Ιούνιο του τρέχοντος υιοθέτησε μια νέα εκδοχή των κατευθυντηρίων γραμμών για τα θέματα σύγκρουση συμφερόντων. Καταρχάς, περιλαμβάνει το θέμα της ε, σύγκρουσης συμφερόντος. Κάθε αντιπροσωπεία πρέπει να συμπληρώσει μία δήλωση των συμφερόντων της από πριν, πριν μπορέσει να αποτελέσει μέλος της αποστολής. Εξακολουθούν να μην υπάρχουν σωστοί ελεγκτικοί μηχανισμοί Πολλέ φορέ κάποια μέλη των αντιπροσωπιών κρύβουν κάποιε πληροφορίε που μπορεί όντω να αποτελούν αντικείμενο σύγκρουση συμφερόντων ή διπλωματία του Χαβιαριού. Και το έχουμε υπογραμμίσει και το μελετούμε πάντα. Τώρα, για τις ε, βέλτιστες πρακτικές Καταρχάς πρέπει να υπάρχει ε, ισορροπία εκπροσώπησης των πολιτικών δυνάμεων. Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό για να εξασφαλίσουμε την αμεροληψία, την ανεξαρτησία της διεθνούς παρατήρησης εκλογών. Οι εμπειρογνώμονε ε, ε, πολιτικών ε, παρατηρήσεων είναι τελείως διαφορετικοί οι εμπειρογνώμονες θα μπορούσε να, μπει κανείς, να πει κανεί για αυτούς. Τους δίνεται αρκετά μεγάλος βαθμός αξιοπιστίας λόγω και των εκθέσεων από τις αποστολές εκλογικής παρατήρησης. Μία από τις βασικές δυνατότητες είναι να δίνεται μόνο μία δήλωση, ε, μία έκθεση μετά τις εκλογές. Να μην υπάρχουν πολλές ή διαφορετικών ειδών από διάφορες οργανώσεις, εκθέσεις, νομοδοτήσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ας πούμε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από τον ΩΣΑ, από την κοινοβουλευτική του συνέλευση. Βεβαίως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις διάφορες απόψεις. Έχουμε την ελευθερία της έκφρασης. Βέβαια, οι πολιτικοί μπορούν να βλέπουν τα πράγματα από διαφορετική οπτική, αλλά ευθύνη των μελών της αντιπροσωπείας είναι να προσπαθήσουν να εξεύρουν μια συμφωνία για την ε, ακριβή διατύπωση, να προσπαθήσουν να συνεργαστούν, ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις όπου η κυβέρνηση παίρνει μια έκθεση παρατηρητών, η αντιπολίτευση παίρνει την άλλη έκθεση των παρατηρητών και δεν υπάρχει κανένα επίπεδο εμπιστοσύνης ή αξιοπιστίας στην, στις εκλογές της χώρας αυτής. Άλλο ένα θέμα λοιπόν είναι και η συνεργασία με τους τοπικούς παρατηρητές που μπορούν να, δώσει, να αποτελέσει μια πραγματική πολύ αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για το τι συμβαίνει ακριβώς στη χώρα αυτή. Η αξιολόγηση των εκλογών είναι μια συνεχής διαδικασία. Δεν ξεκινά τρεις μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών, ούτε τελειώνει την ημέρα που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. Η Επιτροπή της Βενετίας μελετά, όπως είπα, την νομοθεσία σχετικά με τις εκλογές. Οι αποστολές λοιπόν εκλογικής παρατήρησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή, αυτό το πλεονέκτημα της αξιολόγησης του εκλογικού νόμου. Η Επιτροπή της Βενετίας βοηθά καταδεικνύοντας τις ελλείψεις, τα προβλήματα, έτσι ώστε οι εκθέσεις να ε, βασίζονται στην εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής της Βενετίας και η Επιτροπή επίσης μπορεί να αξιολογήσει την νομοθεσία μεταγενέστερα, με βάση τις ε, κακές πρακτικές ας πούμε ή το κατά πόσο η νομοθεσία εφαρμόστηκε καλόπιστα. Και τέλος, στενή συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων και πολιτικών. Είναι και αυτό ένα από τα εχέγγυα της αμεροληψίας και της σωστής αποτελεσματικής παρατηρήσης εκλογών. Βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι όλα τα προβλήματα που αφορούν στις ε, καλές ή τις κακές πρακτικές είναι παρόμοια με, τους, ε, με, τους, με τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα του αθλητισμού, ας πούμε, όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ντόπινγκ και άλλες κακές πρακτικές. Ευχαριστώ κύριε Κάσκ. Μας μιλήσατε ε, για τα όσα ασχολείται η Επιτροπή της Βενετίας. Εγώ έλαβα μία επιστολή πρόσφατα που μου έλεγε πόσο χρήσιμοι είναι οι τοπικοί παρατηρητές μεταξύ των εκλογικών κύκλων, γιατί είναι εκεί στη χώρα, ζουν και μπορούν να έχουν πραγματικές πληροφορίες. Τώρα, να ακούσουμε την ε, κυρία Γκίσλα Ντότυρ. Είναι εκπρόσωπος ε, ε, του γραφείου του ΟΣΑ για, τη, για, για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευθύς εξ αρχής θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας συγκέντρωσε όλους εμάς εδώ από διαφορετικούς φορείς που ασχολούνται με τις εκλογικές παρατηρήσεις. Πολύ θετικό αυτό. Σα ευχαριστώ που με προσκαλέσατε και σε αυτό το πάνελ για τον κώδικα δεντολογία για τι διεθνεί ε, εκλογικέ παρατηρήσει. Για τον κώδικα δεντολογία θα μπορούσα να σα μιλήσω γενικά. Καλό θα ήταν να το εξετάσουμε και από γενική άποψη. Όμως αποφάσισα να επικεντρωθώ σε μία μεμονωμένη πτυχή του κώδικα δοντολογίας, λόγω έλλειψη χρόνου. Πρόκειται για την υποχρέωση διατήρησης, ε, ή μάλλον την υποχρέωση να έχει κανείς μία σωστή προσωπική συμπεριφορά. Στο κώδικα δοντολογίας λοιπόν αναφέρεται ότι οι παρατηρητέ θα πρέπει να συμπεριφέρονται ε, καταλήλως και με σεβασμό προς τους άλλους, να επιδεικνύουν ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα ήθη και έθιμα της ε, χώρας υποδοχής και να διακρίνονται από επαγγελματισμό ε, ανα πάσα στιγμή, ακόμα και στον ελεύθερο τους χρόνο. Όλα αυτά πραγματικά είναι η καρδιά της αξιοπιστίας μας. Πώς μπορεί κανείς να κάνει εξολογήσεις και συστάσεις εάν δεν είναι ο ίδιος ακέραιος και επαγγελματίας. Για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο αποστέλουμε χιλιάδες ε, παρατηρητές σε τέτοιου είδους αποστολές. Πέρσι μόνο είχαμε 2.000 περίπου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το ζήτημα για τον Ότιρ. Εγώ ξεκίνησα πριν από 1,5 χρόνο περίπου, όταν ε, άρχισε να ανεβαίνει η δυναμική του κινήματος Μητού και άρχισε ο κόσμος σιγά σιγά να συνειδητοποιεί πόσο συνήθι φαινόμενο είναι η σεξουαλική παρενόχληση. Ακόμα και στο πλαίσιο των ε, αποστολών παρατήρησης. Αυτό που έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια είναι το επίπεδο ανοχής απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές. Και εμεί πήραμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ακόμα ε, και εκ των προτέρων, να αποτρέψουμε τέτοιου είδους φαινόμενα στο περιβάλλον μας. Πρέπει να ε, εξετάσουμε νέες ιδέες και πρακτικές για το τι είναι αποδεκτή συμπεριφορά και τι όχι. Πρέπει να ακολουθούμε λοιπόν πρακτικές ε, κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης ε, και της διάκρισης με βάση το φύλλο. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο έχουμε υιοθετήσει στο Νότιρ και συμπληρώνει τον κώδικα τεντολογίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο εντάσσεται εδώ και πολλά χρόνια στα εγχειρίδια και στις ε, ενημερώσει που κάνουμε στου παρατηρητέ, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε πραγματικά ενισχύσει σημαντικά τι προσπαθίες μα σε αυτό το πλαίσιο. Προσπαθούμε επίση να ξεκαθαρίσουμε ότι ο οργανισμό μα ακολουθεί μια πολιτική μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση και στο περιβάλλον μας, στα γραφεία μα και στι αποστολέ μα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η ευθύνη μα να διασφαλίσουμε ότι όσοι απασχολούνται από τον οργανισμό μας και όσοι μας αποστέλλονται από τα συμμετέχοντα κράτη και είναι, αλλά και νιώθουν ασφαλείς από τη σεξουαλική παρενόχληση και από οποιαδήποτε άλλη απειλή. Πρέπει να έχουμε λοιπόν κατά νου τις βασικές αρχές της εμπιστευτικότητας και γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πρώτον ε, το θύμα, το, το δυνητικό θύμα μπαίνει στο επίκεντρο της προσέγγισής μας και ότι πρέπει να λάβει την απαραίτητη στήριξη και δεύτερον ότι καλύπτουμε όλο το προσωπικό μας και το εθνικό προσωπικό σε απομακρυσμένες περιοχές και με λιγότερη γνώση, για παράδειγμα, της Αγγλικής. Και τρίτον, ότι ε, δημιουργούμε με διαφορετική νοοτροπία. Πρώτον, επομένως, από πλευράς ε, εξελίξεων τώρα, υπάρχει ένα νέο έντυπο, το οποίο δημοσιεύσαμε, ε, που εμπεριέχει μια σειρά πληροφοριών σε αυτά τα θέματα. Έχουμε φτιάξει και μια αφίσα που χρησιμοποιείται σε όλες τις αποστολές μας για αυτό το θέμα. Έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένες παρουσιάσεις για το επαγγελματικό χώρο εργασίας που παρέχεται σε όλους ε, τους παρατηρητές. Ενισχύουμε ε, την επικοινωνία με τρίτες χώρες τις οποίες στέλνουμε αποστολές και το έχουμε, αναφέρεται αυτό πλέον ρητός στους όρους αναφοράς και τέλος έχουμε ενισχύσει αυτό το σκέλος στις καταρτήσεις που παρέχουμε στα λεγόμενα focal points, σε σημεία εστίαση στα διάφορα συμμετέχοντα κράτη. Έχουμε καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να αλλάξει και η νετροπία και ε, σε ό,τι φορά και του επικεφαλεί των αποστολών. Δηλαδή, ο επικεφαλή αποστολή θα πρέπει να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε αυτό τον τομέα. Και το ίδιο το πρόσωπο αυτό, είτε ένα άντρα είτε γυναίκα, αντιμετωπίζει ε, αποτελεσματικά αυτά τα ζητήματα. Σε όλες τις ε, αποστολέ μα, οι παρατηρητέ πρέπει να υπογράφουν τον κώδικα δεντολογία και αν υπάρχει σοβαρή παράβαση αναφέρεται ότι μπορεί αυτό να οδηγήσει σε άμεση απομάκρυνση της και αφαίρεση της πιστοποίησης. Νομίζω ότι έχω καλύψει τα περισσότερα από τα μέτρα που έχουμε υιοθετήσει για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι υιοθετήσαμε αυτά τα μέτρα γιατί ξέρουμε ότι οι παρατηρητές ότι είναι εκπρόσωποι ε, το, του οργανισμού μας. Είναι λοιπόν και θέμα φήμης για εμάς, υπόλοιψης. Πρέπει λοιπόν να διέπονται και να διακρίνονται από επαγγελματισμό. Ταξιδεύουν σε πολλές ε, τοποθεσίες, ε, συναντούνται με πολλούς αξιωματούχους και εν ώρα και εκτός. Εμείς δεν κάνουμε διάκριση προς αυτό και οποιαδήποτε στάση τους ε, έχει αντίκτυπο και στην, ε, στη φήμη και υπόλοιψη του οργανισμού μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, που αναφερθήκατε σε αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Χαίρομαι, διότι έχουμε 30 λεπτά μπροστά μας στη διάθεσή μας και νέα. Ε, ε, έχουν ζητήσει τον λόγο. Επίσης, δεν θα μιλήσει κανείς πάνω από δύο λεπτά. Εσείς πρώτα και μετά... Ωραία, θα, θα, θα μαζέψουμε όλα τα έντυπα από όσους ζητούν το λόγο. Λοιπόν, το θέμα της ε, καλύτερης παρατήρησης, ελέγχου μάλλον ε, από το ελέγχου των αποστολών από την πλευρά των κοινοβουλίων ε, το οποίο σχετίζεται και με τον κώδικα ε, δεοντολογίας είναι πολύ σημαντικό θέμα. Τον κύριο Βίκτορ Πάους θα ζητήσω τώρα να, α, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τους οργανωτές αυτής της διάσκεψης που έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή, ε, γιατί Πραγματικά ε, και ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, πάρει μέτρα έτσι ώστε να καλυφθούν ζητήματα δεοντολογίας. Υπάρχει και έγγραφο σχετικό με τον κώδικα δεοντολογίας και την ηθική διάσταση της ε, συμμετοχής σε ε, αποστολές παρατήρησης. Εγώ ο ίδιος οποτεδήποτε συμμετείχα σε τέτοιες διαδικασίες ε, μελέτησα προσεκτικά και παρατήρησα τα ζητήματα και έχω καταλήξει ότι υπάρχουν δύο πεδία δυνατότητας βελτίωσης στο μέλλον καταστάσεις ε, οι οποίες ε, κατά την, κατά την άποψή μου ε, αξίζουν συζήτηση Ε, έτσι ώστε ε, να ε, μειωθούν τα ενδεχόμενα προσωπικών συμπεριφορών όχι ικανοποιητικών. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να, να, να θεωρήσουμε σαν ενδεχόμενο την απαγόρευση συμμετοχής, αλλά την δυνατότητα προσθήκης άλλων στοιχείων στον ήδη υπάρχοντα κώδικα δεοντολογίας. Ε, τα θέματα τα οποία θέλω να αναφέρω είναι τα εξής. Περιπτώσεις όπου ε, βουλευτές ως μέλη της Επιτροπής Φιλίας με τη συγκεκριμένη χώρα πηγαίνουν σε εκείνη τη συγκεκριμένη χώρα να, κάνουν παρατήρηση εκλογών. Δεύτερον, περιπτώσεις όπου βουλευτές οι οποίοι ανήκουν ε, σε κόμματα που εκπροσωπούν εθνικές μειονότητες και παρατηρούν εκλογές σε μια χώρα Β, όπου η ε, αναφερόμενη μειονότητα της πρώτης χώρας αποτελεί την ε, πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος ε, τη στιγμή των εκλογών. Πιστεύω ότι δεν είναι ώρα για αποκλεισμούς, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τουλάχιστον δύο ζητήματα. Α, εάν ο βουλευτής την ώρα που υπογράφει τον κώδικα δεοντολογίας ε, ότι ανήκει σε μία από τις δύο κατηγορίες που ανέφερα προηγουμένως, και δεύτερον, για τέτοιες περιπτώσεις μήπως θα έπρεπε να υπάρξουν συγκεκριμένες διατάξεις δέσμευσης ε, που να αναλυφθούν συγκεκριμένα και εν υπογράφος από τους ε, βουλευτές οι οποίοι συμμετέχουν στις ε, εκλογές, ε, στην διαδικασία εκλογικής παρατήρησης. Τελειώνω, τελειώνω. Για να μειωθούν ενδεχόμενες, ενδεχόμενοι πειρασμοί να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Επομένως, ε, τα διάφορα όργανα τα οποία εξειδικεύονται στην παρατήρηση εκλογών θα πρέπει να ε, μελετήσουν τα θέματα, για κυρίως για τις περιπτώσεις που ανέφερα προηγουμένως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναφερθήκατε και στον ρόλο των πολιτικών κομμάτων και των ε, ομάδων φιλίας. Παρακαλώ πολύ συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, λέει η κυρία Γκίλ να αναφερθώ σύντομα σε ορισμένα θέματα σχετικά με τις ελλείψεις που βλέπουμε σε αυτές τις διαδικασίες παρατήρησης και πώς μπορούμε να, τα αντιμετωπίσουμε, να τις αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως υπάρχουν πολλές ε, παρατηρήσεις, αλλά να πω για μια χώρα όπου παρατηρούμε ένα μέλος από μια πολύ ισχυρή χώρα που πήγε εκεί δεν έχουμε κανένα ίχνος, ε, είχε συναντήσεις, επαφές και το βράδυ των εκλογών ε, έκανε ε, μίλησε σε μια συνέντευξη τύπου, έδωσε την άποψή του, την εντύπωση που είχε για τις εκλογές και έφυγε. Μα δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Εάν πραγματικά προέρχεστε από μια πολύ ισχυρή χώρα, ε, τότε ε, πραγματικά ε, εσείς ενδιαφέρετε που τον τύπο, εσείς που έρχεστε από μια τέτοια χώρα. Επομένως θα πρέπει να, υπάρχει κάποιο, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες δεοντολογίας που να είναι δεσμευτικοί για όλους και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε όλα τα κοινοβούλια. Υπάρχουν πρώην υπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί που έχουν την άδεια κατά κάποιο τρόπο το ελεύθερο να κυκλοφορούν παντού ε, και να μιλούν παντού. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ε, Οποιοςδήποτε δεν συμμετέχει σε ε, εκλογές, σε παρατήσεις εκλογών δεν μπορεί να μιλήσει και όσοι συμμετέχουν θα πρέπει να υποβληθούν σε συγκεκριμένη κατάρτιση. Δεύτερη ερώτηση. Πέντε δεύτερα έχεις. όσον αφορά τη χρήση των πόρων. Μερικές φορές, ε, το είπατε και εσείς, ε, ε, μερικές φορές μπορεί κάποιοι να έχουν πικρία και να ε, να, να μην ε, έρχονται σε επαφή και με ε, γηγενείς παρατηρητές. Πρέπει να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των εντός και εκτός. Επίσης, capacity building σε χώρες εταιρική σχέσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι αφήνουμε πίσω μας δηλαδή μετά από την παρατήρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Νίνα, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρομπέρτο Μοντέλα. Γενικό Γραμματέα του, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΑΣΑ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ και την Κριστίνα και εσάς ε, που κάνατε, ε, ε, οργανώσατε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα διάσκεψη όσον αφορά τον κώδικα δεοντολογίας. Και εμείς στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση προσπαθούμε να είμαστε πιο δεσμευτικοί, πιο ισχυροί ε, έτσι ώστε να γίνει ισχυρό και ο κώδικας δεοντολογίας. βεβαίω είναι καλό να υπάρχει ο κώδικας, ίσως μάλιστα και κάποιος κοινό ε, κώδικας ε, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Εγώ ωστόσο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του κοινού σε ένα σημείο. Εδώ και 20 χρόνια παρατηρώ εκλογές και το τελικό προϊόν στο, μετά το πέρασε είναι ένα preliminary statement of conclusions και τελικά μια τελική έκθεση, δηλαδή ένα έγγραφο ε, μερικών σελίδων που δίνεται ε, στο στους εμπλεκομένους 48 ώρες πριν τις εκλογές. Νομίζω πάντως ότι η παρατήρηση εκλογών και ο αντίκτυπος που τα μέλη του Κοινοβουλίου μπορεί να έχουν στο τελικό προϊόν που παράγεται, την τελική έκθεση δηλαδή μετά από την ε, ε, παρατήρηση, ίσως είναι 5-10% μέσα σε ορισμένε περιπτώσεις, ε, γιατί διαπραγματευόμαστε, συζητούμε κτλ. Αλλά ο πραγματικός αντίκτυπος είναι στην ουσία 10 με σε ορισμενε περιπτωσεις γιατι διαπραγματευομαστε συζητουμε κτλ αλλα ο πραγματικος αντικτυπος ειναι στην ουσια 10 Βεβαίως είναι σημαντικό να έχουμε έναν δεσμευτικό κώδικα ε, δεοντολογίας ε, στην ε, κοινοβουλευτική άσκηση των καθηκόντων, αλλά να μην ξεχνάμε το αυτό το 90% που αφορά τον ίδιο τον κόσμο. Το 90% των δηλώσεων γράφεται είτε από τον επικεφαλής, είτε από τον, της αποστολής, είτε από τον αναλυτή εμπειρογνώμονα, από ανθρώπους που είχαν, έχουν και μεγάλη εμπειρία. Μερικοί εξ αυτών βρίσκονται και σήμερα εδώ. και εμείς ε, λέμε ότι θα πρέπει ο κώδικα διοντολογίας να είναι αυστηρό έτσι ώστε να μην υπάρχουν παραστρατήματα, λογοφιλίας ε, κτλ. Άρα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μέσω του κώδικα διοντολογίας αποφεύγονται όλα αυτά. Αλλά και οι εμπειρογνώμονες να όντα είναι, άνθρωποι είναι. Δεν μπορεί να είναι απολύτως ουδέτεροι. Ε, ε, υπάρχουν πολλοί ε, παρατηρητές, διορθώνω πολλοί εμπειρογνώμονες, εκ των οποίων τους γνωρίζω και εγώ, που έχουν βεβαίως σαφείς πολιτικές απόψεις και μάλιστα σαφείς πολιτικές ε, απόψεις για τη χώρα για την ε, οποία καλούνται να συγγράψουν την έκθεση παρατήρησης. Και αυτοί θα πρέπει να υφίστανται κάποιο είδος κώδικα δεοντολογίας. Ε, ξέρουμε ότι για τους βουλευτές ε, ε, υπάρχει ένα θέμα λογοδοσίας. Είπαμε προηγουμένως την, δημο, τη, διπλωματία του Χαβιαριού, αλλά αυτοί αφορούν το 10% της παραγόμενης εργασίας. Το 90% της εργασίας που παράγεται μέσω της έκθεσης και αυτά γίνεται από τους εμπειρογνώμους και αυτά. Άρα, άρα και, και εδώ παρακαλώ να μην θεωρήσετε ότι κατηγορώ οποιονδήποτε. Δεν θέλω να ε, γίνω πολέμιος ε, κάποιων κατηγοριών, ας πούμε, εμπειρογνωμών κτλ. Αλλά είναι και αυτοί οι ανθρώπινα όντα, δεν είναι ουδέτεροι Άρα θα πρέπει, εάν θέλουμε πραγματικά να είναι ε, ακέραιοι και ανεξάρτητη η εργασία, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και αυτοί που παράγουν το 90% της εργασίας και της τελικής έκθεσης. Άρα θα πρέπει ε, να είμαστε και σίγουροι ότι ο μηχανισμός πρόσληψης αυτού του 90% ε, ε, είναι σωστός. Προφανώς το θέμα αφορά αυτούς που έχουν τις ευθύνες. Ναι, δυστυχώς πρέπει να δώσω το λόγο στην κυρία μας, της Βελγικής Συγκλήτου. Um, former and current MPs. Κάποιοι από τους ευρωβουλευτές μας ασχολήθηκαν με μια βελγική περίπτωση και δεν είναι πλέον καλοδεχούμενοι στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Σε εθνικό επίπεδο κάναμε μια συζήτηση για το ποιες είναι οι πιθανές κυρώσεις που θα μπορούσαν να υπάρξουν σε εθνικό επίπεδο για τα άτομα αυτά και δεν ήταν τελικό σαφές τι θα γινόταν. Ήταν δύσκολο λοιπόν αυτό. Ερώτημα προς όλους, αλλά κυρίως προς τον ΩΣΑ μπορείτε να, μπορούμε, μπορείτε να αρνηθείτε αυτά τα άτομα να πάρουν μέρος σε μελλοντικέ αποστολές ε, με βάση εκθέσεων άλλων οργανώσεων, με βάση εκθέσεις άλλων οργανώσεων ή πρέπει να έχετε την άδεια ας πούμε, του εθνικού επίπεδου για να το κάνετε αυτό. Τι προτείνετε. Άκουσα ότι προτείνετε να εφαρμοστεί ο ίδιος κώδικας δεοντολογίας σε εθνικό επίπεδο. Είναι ρεαλιστικό αυτό. Είναι εφικτό. Πώς μπορείτε να το κάνετε. Γιατί θέλουμε να αποφύγουμε άτομα που έχουν όντως ε, συμπεριφερθεί με ανάρμοστο τρόπο, προφανέστατα να μην μπορούν να πάνε σε μελλοντικέ ε, διεθνεί ε, τέτοιε αποστολέ. Οπότε εσείς τι προτείνετε για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Μάς. Χωσέ επόμενος ο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε συνάδελφο Ευρωβουλευτή. Ναι, Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να τηρήσω και το όριο των δύο λεπτών. Okay, great. Sorry, wrong Michael. Um, I'll try to skip to the two minutes. Um, Antes de mais, quero agradecer a, participação dos palestrantes, especialmente da doutora Isabel Santos e da senhora Gisla Dottir. Καταρχικά να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, ιδίως τους δύο πρώτους. Ε, συμμετείχα σε πολλές από τις αποστολές εκλογικής παρατήρησης ως μέλος ε, των κοινοβουλευτικών επιτροπών που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το έργο και πολύ σημαντικά τα όσα είπατε και συμφωνώ. Και εγώ πρόσφατα μάλιστα πήγα στο Μαυροβούνιο σε τέτοια αποστολή Και εμείς είχαμε μια τέτοια περίπτωση όπου ένας συνάδελφος ε, αποκλείστηκε από την αποστολή. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Όμως απλώς θέλω να πω ότι ήμουν μάρτυρας αυτής της ε, κατάστασης. Τώρα, να αναφερθώ σε κάτι πολύ σοβαρό που μπορεί να λάβει η χώρα εκτός της ε, αποστολής αυτής. Να σας δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Σε μια εκλογική αναμέτρηση εντός αγωγικών προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα. Οι συνάδελφοι στην οποία αναφέρθηκε η πρόεδρος της ΟΤΙΡ ε, ήταν ε, ε, το πρόσωπο του θεσμικού αυτού οργάνου. Τι γίνεται με την υπόλοιψη ενός αυτού του οργανισμού. Ένας ή δύο συνάδελφοι συμμετείχαν εκεί χωρίς να έχουν λάβει εντολή και άδεια. Και είδαμε στα κοινωνικά δίκτυα τι κυκλοφόρησε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε αυτούς τους βουλευτές. Και να αναφέρω και κάτι άλλο. Όταν εξετάζουμε αυτό το ζήτημα και σε σχέση με τη συμμετοχή των ε, ε, βουλευτών πέραν των πλαισίων της ε, αποστολής, έχετε δίκιο ότι αυτός ο κώδικας συντολογίας θα πρέπει να ισχύει για όλους. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβλέπετε ο κώδικας οντολογίας για όλους τους βουλευτές που προσκαλούνται και από τις ε, τοπικές αρχές, για παράδειγμα. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Thank you, colleague uh, Faria. And the next... Ευχαριστώ. Λένα Σινάιπ από την Ομοσπονδία των Αραβικών Κρατών, η επόμενη ομιλήτρια. Actually, uh, I didn't. Uh, ah. Did you say you did not ask for the floor? Δεν ζητήσατε το λόγο. Α, συγγνώμη. Νικολάη Πάνφελ από την Πόμολεξ από την Μολδαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα του σημερινού πάνελ είναι οι καλές πρακτικές για την παρατήρηση εκλογών. Θα ήθελα να μιλήσω από την ε, πλευρά των, του εκπροσώπου των ε, οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών που κάνουμε σε τοπικό επίπεδο τέτοια παρατήρηση και πραγματικά ε, θα πρέπει οι διεθνεί οργανισμοί να έχουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία σε τοπικό επίπεδο με του τοπικούς, του ντόπιου ε, παρατηρητές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορώ να σας μιλήσω για την κατάσταση που είχαμε, ας πούμε, το 2009, όταν έγινε αυτή η επανάσταση στο Twitter και τι είδους επικοινωνία υπήρχε μεταξύ των διεθνών και των ντόπιων παρατηρητών, αλλά και ποιες είναι οι συνέπειες που είχαμε στη χώρα μετά από αυτό είχαμε ε, εκλογές τον Απρίλιο. Και τα τελευταία χρόνια η επικοινωνία αυτή έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Και αυτό πραγματικά έχει ωφέλη και για τους ντόπιου παρατηρητές, των οποίων τα ευρήματα και οι συστάσεις ε, λαμβάνονται υπόψη και φτάνουν στα ανώτατα επίπεδα, αλλά και οι δικές σας οι εκθέσεις γίνονται πιο συνεκτικές γιατί εμείς έχουμε τις επιτόπου πληροφορίες και μπορούμε να καλύψουμε πολύ μεγαλύτερες περιόδους παρατήρησης. Επίσης, θα ήθελα να σας καλέσω στα πλαίσια των επόμενων βουλευτικών εκλογών τον Φεβρουάριο στην, στην Μολδαβία να δώσετε προσοχή στην εφαρμογή ή στην προετοιμασία αυτών των εκλογών στα πλαίσια Τη εφαρμογής της μεταρρύθμισης του εκλογικού συστήματος που έγινε πρόσφατα. Η μεταρρύθμιση αυτή δεν έγινε με πολύ διαφανή τρόπο και με καθόλου συμμετοχικό τρόπο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω και επίσης θα ήθελα να σας καλέσω μια που οι τοπικές οργανώσεις δεσμεύονται από κώδικα δαντολογίας εμείς έχουμε πολλούς εμπειρογνώμονε, πολλούς ειδικού που δουλεύουν στις διάφορες χώρες, σε διάφορες οργανώσεις και οργανισμούς. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο είδος συνεργασία, όχι κατά τη διάρκεια μόνο τη ε, ε επικοινωνία στη χώρα, όταν δηλαδή συναντιόμαστε, αλλά θα μπορούσαμε ίσω να, να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό ώστε να γίνουμε και εμείς ε, μέλη διεθνών αποστολών για να μπορέσουμε να, να, να ανταλλάξουμε πληροφορίες έτσι ώστε να υπάρχουν στην ομάδα αυτή ε, και οι δύο απόψεις. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, όλοι γνωρίζουμε το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με την ε, κοινωνία των πολιτών και με τις οργανώσεις της. Έχω τρεις ομιλητές ακόμη. Θα τους ακούσουμε και μετά θα επανέλθουμε στο πάνελ. Ο κύριος Μάθιου Σάλιγκ από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Πολύ σύντομη θα είναι η δική μου παρέμβαση, Πρόεδρε. Δύο, ερώτημα έχω για, δύο ερωτήματα έχω για τους ε, πανελίστες. Με τον νέο κώδικα δοντολογίας, σε ποιο βαθμό οι οργανώσεις σας θα δώσουν ε, κατάρτιση και θα κάτσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι με τους ε, κοινοβουλευτικούς για να τους εξηγήσουν ποια είναι τα σημαντικά θέματα και ε, ποια είναι τα προβλήματα εάν δεν τον τηρήσουν. Και επίσης, σε ποιο βαθμό θέλετε να ενισχύσετε τους αναπληρωτές ή τους επικεφαλείς που συνοδεύουν τους κοινοβουλευτικούς παρατηρητές για να εφαρμόσουν τον κώδικα δοντολογίας. για να, το, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν συμβαίνει και όχι όταν έχει γίνει η ζημιά εκ των υστέρων. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Σάλικ. Στέφανη Σίφερ από την EPD. E. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ ένα δίκτυο 40 οργανώσεων στην Ευρώπη και θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για τον νέο κώδικα τοντολογίας που είναι πολύ θετικό βήμα. Περιλαμβάνει και συστάσεις που προκύπτουν από ε, τέτοιους οργανισμούς εκλογικών αποστολών. Είναι όμως το πρώτο βήμα, όχι το τελευταίο. Το επόμενο βήμα ποιο πρέπει να είναι. Τα εθνικά κοινοβούλια ε, στην Ευρώπη να υιοθετήσουν τέτοιους κώδικες δεντολογίας. Το αναφέρθηκε προηγουμένως. Και να σας πω γιατί είναι τόσο σημαντικό. Στις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία τον, ε, το υπήρχε μια μεγάλη έκθεση που όμως δεν άκουσαν οι ε, Ρώσοι πολίτες ε, τα πορίσματα αυτής της έκθεσης. Άκουσαν όμως ε, τους 400 και πάνω απεσταλμένους από, από ευρωπαϊκές χώρες που είχαν προσκληθεί από την Ρωσία παρευρέθησαν μόνο την ημέρα της, των εκλογών και δεν παρουσίασαν κάποια ε, επίσημη έκθεση, αλλά ε, ουσιαστικά μετέφεραν θετική εικόνα και έτσι επισκίασαν ε, τις παρατηρήσεις ε, της αποστολής. Κάτι αντίστοιχο έχουμε δει και στη Ζιμπάμπουε. Υπήρχε μια αποστολή 32 ατόμων στην Καμπότζη. Ήθελα λοιπόν να πω ότι αν οι διεθνείς οργανισμοί ε, αυξήσουν και ενισχύσουν τους κώδικες εντολογίας, το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Thank you very much for this uh, observation. Ευχαριστούμε, Στεφανή. Τελευταίος ομιλητής. Τελευταίος. Γκάιλ Μάρτιν Ντικαλέ από την Επιτροπή της Βενετίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χάουταλα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το, το Γκαέλ συχνά το περνάνε για γυναική όνομα, δεν, δεν με ενοχλεί. Ένα σύντομο σχόλιο και μετά ένα ερώτημα. Αρχικά όλοι θα συμφωνήσετε ότι είτε πρόκειται για εκλογικούς ε, παρατηρητές ε, πολιτικοποιημένους ή μη, ή τεχνικούς ε, παρατηρητές, είτε πρόκειται για πολιτικούς ε, παρατηρητές, όπως εδώ οι βουλευτές για παράδειγμα, στο πλαίσιο των διεθνών αποστολών εκλογικής παρατήρησης, που συχνά είναι και του ΝΑΤΟ, του ΟΣΑ, του Ευρωκοινοβουλίου βεβαίω και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο συζήτησα και με συναδέλφους που δεν μπορούσαν να είναι εδώ σήμερα γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται και μία ε, σύνοδος ε, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στο Στρασβούργο. Απλώς θέλω να σας μεταφέρω το μήνυμα ότι σε ό,τι φορά και τις ε, γενικές ε, αρχές που υπεγράφησαν το 2005 στο πλαίσιο του ΟΗΕ, αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις στο Αζερβαϊτζάν και προβλήματα διαφθοράς με συγκεκριμένους βουλευτές. Η ε, Κοινοβουλευτική Σύνοδος, λοιπόν, ενίσχυσε και κατέστησε πιο αυστηρές τις καθημερινές γραμμές, αλλά και την δήλωση συμφερόντων των υποψηφίων που πρέπει να υπογράψουν όλοι οι βουλευτές. Πρόκειται και μια δήλωση βεβαίως, Επομένω, προποθέτει και την ειλικρίνεια και την ε, ηθική ε, του ε, εμπλεκομένου, αλλά επανέρχομαι στον κώδικα δεντολογίας που θα υιοθετηθεί και θα εφαρμοστεί από τις διάφορες αποστολές, θα πρέπει να καθιστά υποχρεωτική την υποβολή αποδείξεων σε ό,τι αφορά το ήθους και την ανεξαρτησία των συμμετεχόντων. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα πρέπει να αυτοσχεδιάσω, γιατί βλέπω ότι πολλά μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, γιατί δεν μπορούν να πάρουν το λόγο. Αλλά δέχεστε να πάρετε το λόγο, αλλά για ένα λεπτό. Λυπάμαι, αλλά ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος from ε, the Romania. Ο κύριος Ρωμασκάνο από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 37 δευτερόλεπτα. Θα μιλήσω εξ ονόματος ε, της Ρωμανικής Εθνικής Αντιπροσωπείας των OACPA. Με περηφάνεια μπορούμε να σας πούμε ότι από την αρχή της, ε, του εγχειρήματο της παρακολούθησης της παρατήρησης εκλογών συμμετείχε η Ρουμανία με δύο βουλευτές το 1993 για το δημοψήφισμα στη Ρωσία το 1993. Μόνο ένα σημείο ήθελα να Βλέπουμε ότι πολλέ ευρωπαϊκέ οργανώσει ασχολούνται με την παρατήρηση εκλογών. Ίσως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο λοιπόν δημιουργία μια διακοινοβουλευτική ομάδα με μέλη του SCPA, του Συμβουλίου τη Ευρώπη, ε, του ΝΑΤΟ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχουν και ηγούνται τέτοιων αποστολών, με βασικό στόχο την ανάλυση ε, και ανάδειξη ε, ισχυρών στοιχείων και αδυναμιών, τη βελτίωση, των, μάλλον την ενίσχυση των βέλτιστων πρακτικών και την εξέβρεση λύσεων στα πιθανά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις ε, εκλογές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Δίνω το υπόλοιπο του χρόνου μου στο συνάδελφο από τη Σουηδία. Um, Ευχαριστούμε. Μαργαρέτα Σερέκα από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να πω το εξή. Πολλοί παρατηρητέ έχουν ε, δικό, δικούς τους πολιτικούς στόχους Καλό ο κώδικας εντολογίας, καλές οι δηλώσει συμφερόντων, οι ενημερώσεις, εκπαιδεύσει, πολύ καλά όλα αυτά. Όμως, όταν επιστρέφουν στη βάση τους, παρόλα αυτά έχουν δικές τους πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν τους ενδιαφέρει η επίσημη αποστολή. Γιατί και εγώ έχω συμμετάσχει σε τέτοιου είδου αποστολέ και βλέπω ότι είναι ένα εντυνόμενο πρόβλημα. Πρέπει να το έχουμε κατά νου. Φυσικά δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε έναν ε, πολιτικό να εκφέρει γνώμη, αλλά όταν κάποιος συμμετέχει σε μία ε, αποστολή παρατήρησης, θα πρέπει να ακολουθεί ε, την έκθεση. Είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση του προβλήματος, γιατί συχνά πρόκειται για λαϊκιστές. Ή άτομα που έχουν να κάνουν με την απάτη, τη διαφθορά. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Um, Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαρία Τελερίτη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, παρακαλώ. One minute. Με σήματα. Ε... Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, μπορείτε. Ε... Je voudrais poser certaines questions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 Το δεύτερο που θα ήθελα να, να θέσω είναι ένα, ε, όχι ακριβώς ερώτημα, αλλά μια πρόταση που αφορά ε, την ε, συμμετοχή των γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά και των άλλων ομάδων που βιώνει, να βιώσουν κοινωνικό αποκλεισμό. Θα πρέπει εδώ να υιοθετηθεί μια οπτική και στη μεθοδολογία και στα εργαλεία, έτσι ώστε να αποτυπώνονται αυτές οι παρατηρήσεις και η εμπειρία μέσα από την εκλογική διαδικασία γιατί θα πρέπει να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν το σύνολο αυτής της ποικιλομορφία και της διαφορετικότητας του εκλογικού σώματος. Ε, επίσης αυτό θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να μπορεί να αναφέρεται ε, στην τελική έκθεση για να μπορούμε να δούμε πραγματικά τις ε, συμμετοχικές διαδικασίες, την προέλευση δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στην εκλογική διαδικασία αυτών των ομάδων. Και τέλος, πώς διασφαλίζεται με, με την χρήση των τεχνολογιών στην εκλογική διαδικασία η καθολικότητα, η ισότητα και η μυστικότητα της ψηφοφορία, καθώς και η προσβασιμότητα και η διαφάνεια ε, εδώ θα πρέπει να δούμε πάλι τις προδιαγραφές που έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και να τις εμπλουτίσουμε έτσι ώστε να είναι πιο σαφή σε εμά όταν είμαστε παρατηρητές στις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. you ε, Σας ευχαριστούμε. Τώρα ας στραφούμε στους ε, ομιλητές μας, στους τέσσερις οι Να αντιστρέψουμε τη σειρά αυτή τη φορά. Ίγκεμπορκ, θα ήθελες να κάνεις ορισμένες παρατηρήσεις αλλά παρακαλώ να μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά έκαστος. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση. Σε πολλά ζητήματα θα μπορούσα να σταθώ στην τελική μου εδώ παρέμβαση. Θα ήθελα αρχικά να πω ότι όπως ξέρετε ε, είχα αυτή την δυτή ιδιότητα, καθώς ήμουν πολιτικός για πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα είμαι διευθύντρια του ΟΤΙΡ και προσλαμβάνω επαγγελματίες που ασχολούνται στις, ε, με τις αποστολές ε, παρατήρησης. Οπότε κατανοώ και τις δύο πλευρές. Ξέρω ότι οι πολιτικοί πάντα έχουν ε, πολιτικούς σκοπούς, πολιτική ατζέντα, μα είναι φυσιολογικό, γι' αυτό ασχολούνται με την πολιτική. Όμως, όταν συμμετέχουν σε αποστολές στο πλαίσιο μιας ομάδας που καταλήγει σε κοινά συμπεράσματα, είναι πολύ σημαντικό ε, όταν τοποθετούνται να το κάνουν για να προβάλλουν τα συμπεράσματα της ομάδας. Βέβαια δεν μπορούμε να τους απαγορεύσουμε και να τους εμποδίσουμε όταν επιστρέφουν στη βάση τους να παρουσιάζουν διαφορετικά τα συμπεράσματα. Αλλά δεν μπορούν να αντιφάσκουν σε σχέση με την έκθεση. Μπορούν να την ερμηνεύουν με βάση ε, τις δικές τους πεπιθήσεις, αλλά όχι να αντιφάσκουν ως προς αυτήν. Γιατί τότε υπονομεύουν το έργο όλης της αποστολής. Και αυτό δεν ε, μπορεί να γίνει ανεκτό. Είναι δύσκολο να το ε, σταματήσουμε σαν φαινόμενο. Να επανέλθω στα όσα είπε ο Ρομπέρτο για την ε, λογοδοσία, την πολιτική ευθύνη των πολιτικών και των βουλευτών. Πράγματι, οι ε, βουλευτές λογοδοτούν στους ψηφοφόρους τους. Αλλά όταν συμμετέχει κανείς σε μια διεθνή αποστολή, δεν υπάρχει και τόσο λογοδοσία έναντι των ψηφοφόρων. Πηγαίνει κανείς μόνος του με, με τη δική του πολιτική ατζέντα δεν ε, λογοδοτεί ενώπιον των ψηφοφόρων, δεν κατεβαίνει σε κάποιες εκλογές στην πατρίδα του. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εφαρμόζεται ο κώδικας διοντολογίας για όλους. Και μετά για το προσωπικό αυτής της ε, ομάδα. Όταν μιλούσα προηγουμένως στην τοποθέτησή μου, δεν μιλούσα μόνο για, για το επιτελείο, για το προσωπικό μας, αλλά για όλους. Εγώ μπορώ να σα μιλήσω βέβαια για το προσωπικό του Ότιρ και πώ χρησιμοποιούν τον κώδικα εκεί. Αλλά φυσικά και το προσωπικό υπάλληλή μα δεν είναι τελείω ουδέτεροι. Κανεί δεν είναι τελείω ουδέτερο. Όλοι έχουμε τι απόψει μα και πεπιθήσει μα. Όμω, τουλάχιστον εγώ τι ζητώ από του υπαλλήλου μα. Να ε, διακρίνονται από επαγγελματισμό. Να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, να είναι αμερόληπτοι. Και αυτό εγώ μπορώ μόνο να λάβω υπόψη. Αυτό είναι ο ρόλο μου πρέπει να είναι επαγγελματίες. Δεν απαιτώ να μην έχουν γνώμη, αλλά πρέπει να είναι επαγγελματίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ingeborg. Oliver Kask. Εσείς τι αποκομίσατε από τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Πολλές ε, αξιόλογες παρατηρήσεις ακούστηκαν σήμερα. Ένα από τα ζητήματα που γύρεται ήταν αυτό ενός πολιτικού ή ενός εξέχοντος προσώπου που ε, πηγαίνει μετά και παρουσιάζει τη δική του προσωπική γνώμη που αποκλίνει από την ε, έκθεση της ε, Διεθνούς Αποστολής. Λίγα είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Ιδίω τώρα που είναι τόσο διαδομένα τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Πρώτον, είναι μια ευκαιρία για τα εγχώρια μέσα ενημέρωση ή για τις ε, τοπικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει. Πρέπει να αναδείξουν ε, τέτοια περιστατικά. Όταν τα θίγουν και οι επίσημες ε, αποστολές. καθήκον ε, των αποστολών εκλογικής παρατήρησης δεν είναι μόνο να επισημαίνουν ε, τα βασικά πορίσματα της ε, έκθεσης. Σκοπός της αποστολής είναι κάπως να είναι μια χείρα βοηθείας προς τους ε, φορείς διεξαγωγής των εκλογών ή προς τα δικαστήρια που πρέπει να αποφασίσουν σε ό,τι φορά συγκεκριμένε ενστάσεις, για παράδειγμα, για την εκλογική διαδικασία. Εάν λοιπόν υπάρχει μια επίσημη δήλωση, ακόμα κι αν κάποιοι μεμονωμένοι πολιτικοί αποκλίνουν από αυτό το μήνυμα, Ακόμα και αν λένε ας πούμε, ότι όλα έχουν γίνει σωστά στην εκλογική αναμέτρηση, ενώ στην πράξη δεν ισχύει αυτό, πάντα είναι καλό για τους φορείς ε, διαχείρισης των εκλογών ή για τα δικαστήρια να βασίζουν τις εκτιμήσεις τους στα πορίσματα των αποστολών, των διεθνών αποστολών. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι η ανάρμοστη συμπεριφορά ορισμένων προσώπων ή πολιτικές δηλώσεις ατόμων που δεν είναι πολιτικοί ούτε εκπροσωπούν κάποια κοινοβουλευτική ε, σύνοδο. Εκεί το ζήτημα του κώδικα δεντολογίας η πολιτική τοποθέτηση εμπειρογνωμόνων, για παράδειγμα, δεν είναι δεν έχει την ίδια σημασία όσο έχουν τα βασικά έγγραφα που εκπονεί αυτή η αποστολή. Συλλογικά δηλαδή, όχι ένας και μόνο. Συλλογικά εκπονείται ένα έγγραφο ε, στο οποίο αντανακλώνται και διαφορετικές απόψεις. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πώς σας φαίνεται. Ο Μαλτέζος συνάδελφος θα πάρει τώρα τον λόγο. Ο κύριος Γκαλέα. Παρακαλώ, τι γνώμη έχετε εσείς. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Εγώ θα ήθελα αυτός ο κώδικας συντολογίας να είναι υποχρεωτικός. Ιδάλλως, ε, χάσιμο χρόνο πρέπει να είναι δεσμευτικό. Ιδίω ό,τι αφορά του εμπειρογνώμονε, του εκλογικού εμπειρογνώμονε. Εγώ γνωρίζω πολλού τέτοιου εκλογικού εμπειρογνώμονε που είναι επαγγελματίε, αμερόληπτοι. Έχω μάθει πολλά από αυτού, αλλά επιμένω. Θεωρώ ότι θα πρέπει ο κώδικα να είναι υποχρεωτικό και να δεσμεύει του πάντε. Προτείνω επίση τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που να επιβλέπουν και να ελέγχουν τη συμπεριφορά και τη στάση των βουλευτών που συμμετέχουν σε διεθνείς αποστολές. Και να υπάρχει και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση της συμπεριφοράς. Ο Μάτιου Σαλίκ έθεσε ένα ερώτημα. Θεωρώ ότι ο επικεφαλής της επιστολής, αποστολής ε, έχει αυτή την ευθύνη να εξηγεί τον κώδικα τεντολογίας και να μεριμνά ούτω ώστε ε, όλοι οι συμμετέχοντες να τον υπογράψουν και να τον τηρούν. Και πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, αποκλεισμού ενός ε, μέλους από την αποστολή εάν επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι αποστολές με τα πορίσματά τους και είναι σημαντικό να ε, υπάρχει και σωστή επικοινωνία των πορισμάτων προς τα τελικά ενδιαφέρομενα μέρη, αλλά τελικά οι εκλογές δεν ανήκουν σε εμά, ανήκουν στο λαό. Ο λαός ε, είναι το πιο σημαντικό ενδιαφέρομενο μέρος εδώ. Θα πρέπει λοιπόν τα συμπεράσματα και τα πορίσματα να φτάνουν μέχρι το λαό. τι γίνεται μετά το πέρας της αποστολής. Και ο Μάθιο και η Χάνα και η Μαρία τα γνωρίζουν. Ε, στην περιφέρεια των Βρετανικών νήσων και της Μεσογείου, εμείς τι κάναμε, ήταν υποχρεωτικό για τους συμμετέχοντες. Μετά το πέρας της αποστολής, αν θέλουν να δώσουν συνέντευξη ή να σχολιάσουν την εκλογική αναμέτρηση, θα πρέπει να λάβουν την έγκριση του επικεφαλής της αποστολής από πριν. Δεν υπάρχει λοιπόν λευκή επιταγή προς όλους. Αποστέλλεται στον επικεφαλής ε, της αποστολής, ε, λαμβάνουν την σύμφωνη γνώμη και μετά. Ε, ισότητα μεταξύ των φίλων. Αυτό εντάξει, σαφώς και είναι απόλυτη προτεραιότητα. Δεν γίνεται εμεί να δεχόμαστε τέτοιου είδου πρακτικές. Έτσι κι αλλιώ και με βάση και τι συμβάσεις συμβάσει υπάρχει η απαγόρευση οποιασδήποτε διάκριση με βάση τον φίλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια των αποστολών μας. Είναι σημαντικό λοιπόν η ομάδα παρατήρησης να σέβεται την ισότητα των φίλων. Δεν μπορώ... Ή μάλλον είναι σαφής η σημασία ε, του συντονισμού με τις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κάτι τελευταίο, κλείνοντας. Σύγκρουση συμφερόντων και αμεροληψία οι εκλογές κερδίζονται με το συνέστημα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Πάντα ανάβουν τα αίματα αν θέλετε στις εκλογές και ως παρατηρητές πρέπει εμείς φυσικά να είμαστε συναισθηματικά εκεί, αλλά να μην εμπλεκόμεθα. Τέλος, η κυρία Σάντος. Uh, Αντιπρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΑΣΕ. Και παρακαλώ πολύ επειδή αναμένουμε την κυρία Μογκερίνη. Λοιπόν, από τη στιγμή που μπορώ να μιλήσω πορτογαλικά γιατί έχω διερμηνία, ε, θα μιλήσω στη γλώσσα. First, Ήρθαμε όλοι εδώ έτσι ώστε να συζητήσουμε ε, για θέματα που μας απασχολούν όλους, γιατί όλοι έχουμε ζήσει τέτοιες περιπτώσεις, ε, ε, εννοώ αποστολές εκλογών κλπ. Και είναι εξαιρετικά ε, σημαντικό να μιλήσουμε για τις εκθέσεις. Εκθέσεις οι οποίες αποτελούν το επιστέγασμα κατά κάποιο τρόπο των αποστολών. Ωστόσο, να μην λησμονούμε ότι ε, αυτές τις εκθέσεις τις εκπονούν ε, συγκεκριμένοι οργανισμοί ε, και δεν αναφερόμαστε και σε παράλληλες αποστολές, ενώ είναι όλο και περισσότερες οι παράλληλες αποστολές. E eh, και οπωσδήποτε ε, είναι γεγονός ε, ωστόσο ότι οι εκθέσεις ε, των αποστολών και οι γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται όλο και περισσότερο υπόψη. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Γιατί διαφορετικά, γιατί να τα κάναμε όλα αυτά και γιατί οι κυβερνήσεις να έστελναν παράλληλες ας πούμε αποστολές. Θα χρηματοδοτούσαν μονάχα ε, κάποιες ε, παράλληλες αποστολές τις οποίες θα είχαν προκαλέσει οι ίδιοι έτσι ώστε να μιλήσουν με καλά λόγια για τους πολιτικούς ε, στη συγκεκριμένη χώρα. Ε, από τη στιγμή που υπάρχουν όμως ε, άνθρωποι οι οποίοι ε, εκφράζουν την αποψή τους, τους οποίους ακούν οι πάντες, καταλαβαίνουμε, άλλωστε μιλισμονούμε ότι είμαστε όλοι παρόντες στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, στα tweets, στα Facebook, στα διάφορα. Και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό ο, ο καθένας από τους βουλευτές όταν λέει ότι πρέπει να ενδυναμωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης να ελέγχει πρώτα ο ίδιος τον εαυτό του. Νομίζω ότι οι πολιτικοί και οι βουλευτές ε, γνωρίζουν τις διαδικασίες, ε, έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, έχουν τις απαραίτητες, ε, ε, τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεδηλωμένες πολιτικές απόψεις, άρα μπορούν ανα πάσα στιγμή να ελεγχθούν όσον αφορά ε, την ανεξαρτησία των λόγων τους. Βεβαίως πάντα μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν κάποιοι ε, οι οποίοι να μην κάνουν καλά τη δουλειά τους φυσικά και από την άλλη πλευρά ε, είναι γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να έχει κάποιες δικές του προσωπικές απόψεις ή κάποιες δικές του προσωπικές επιθυμίες. Ωστόσο, αυτές θα πρέπει να τις βάλει κατά μέρος και θα πρέπει να αναφέρεται μονάχα στα πραγματικά περιστατικά, σε αυτά τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της παρατήρησης των εκλογών και επομένως η τελική έκθεση να είναι όσο γίνεται πιο αντικειμενική και πιο διαφανής. Το θέμα των γυναικών επίσης ε, είναι πολύ σημαντικό. Ε, ε, επανειλημμένα έχουμε επιστήσει την προσοχή στο γεγονός της μειωμένης συμμετοχής γυναικών και στο γεγονός ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε τέτοιου είδους αποστολές. Επίσης να αυξηθεί και η παρουσία των γυναικών στους εκλογικούς καταλόγους ε, στις εκλογικές ε, λίστες, τα ψηφοδέλτια. Αυτά ήθελα να σας πω και δεν, θέλω να ε, πω τίποτα παραπάνω. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, δικές σας παρατηρήσεις. Θα κάνω μια εξαιρετικά σύντομη τελική παρέμβαση εν είδη τελικού συμπεράσματος, γιατί νομίζω ότι όλοι εμείς που είμαστε εδώ γνωρίζουμε πόσο σημαντικό εργαλείο είναι ακριβώς αυτό το εργαλείο της παρατήρησης εκλογών. Διαπιστώνω πάντως ότι πρέπει να ε, εφαρμοστεί ο κανόνας ε, δεοντολογίας ε, και μάλιστα μερικοί είπαν ότι ίσως θα πρέπει να υπάρχει κοινό κώδικας δεοντολογίας για τις, για τις τέσσερις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν ή θα έχουν ένα τέτοιο κώδικα. Πραγματικά αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ε, μια συνεδρίαση, ε, τέτοια διάσκεψη ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με παρόμοιο αντικείμενο. Ωραία, τώρα Τώρα θα ήθελα απλώς να σας πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που ολοκληρώσαμε και αυτή τη συνεδρίαση και να σας παρακαλέσω να παραμείνετε στην αίθουσα γιατί είπα ότι εκπρόσωπος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρία Μαργαρίτα Μπογκερίνη θα είναι εδώ μαζί μας σε λίγο.